Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει και πάλι η συνεδρίαση. Έχετε τα πρακτικά της θεσινής συνεδρίασης ε, στην διάθεσή σας. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα θεωρήσω ότι έχουν εγκριθεί. Περνούμε στο πρώτο σημείο μας, κοινή συζήτηση που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Έχουμε πρώτα απ' την έκθεση του κυρίου Ζουβά για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και δύο εκθέσεις του κυρίου Ταραμπέλα για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στο τομείς ύδατο, ενέργεια, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Δεν μπορεί να είναι σήμερα το απόγευμα εδώ ο κύριο Ζούδα και θα αντικατασταθεί από την κυρία, την συνάδελφό του, Τούρμουν Χόφελστάιν. Η κυρία συνάδελφος Τούνουν Χόχανστάιν έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο συγητής δεν μπόρεσε να παρευρεθεί όπως ακούσαμε. Ζητήσει συγγνώμη για την απουσία του.